πάνω από οποιοδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντόλ και τώρα το λόγο στον κύριο Μάρτιν Σούλς για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Σπάνια σπάνιστερη περιπτώσει όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε να συζητήσει προετοιμασία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συνθήκε χειρότερε από αυτέ τη τωρινή κρίση και νομίζω ότι δεν έχει κανεί ψευδεστήσει πλέον. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό έχει ιστορική σημασία. Ιστορική σημασία γιατί λαμβάνει αποφάσει και για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την εβδομάδα διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον ε, ε, χωρίο σε μια, ευρωπαϊκή, σε μια γερμανική ε, εφημερίδα όπου έλεγε στο άρθρο ότι ο Ευρωπαίος πολίτης δυσπιστεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν τη έχει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματά του. Ο πολίτης στην Ευρώπη δυσπιστεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματά του. Είμαστε μέσα σε μια βαθιά κρίση, σε μια κρίση πάνω απ' όλα εμπιστοσύνης για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Είναι γνωστά τα προβλήματα, Έχουμε όλη αυτή την κόπωση από την κρίση. Από την κρίση. Το θέμα είναι αν μπορούμε να δώσουμε τα σκληρά, σκληρές απαντήσεις που Αν Έχουμε το θάρρος και την παρησία να τις ε, προβάλλουμε αυτές τις απαντήσεις ή αν από, από αδράνεια θα, θα αφήσουμε τις εξελίξεις να μας ξεπεράσουν. Και θα ήθελα να πω γιατί το πιστεύω βαθύτατα ότι αυτό θα μας βάλει από την κρίση, ότι από αυτές τις συνθήκες δεν χρειαζόμαστε λιγότερη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε το θάρρος και την παρησία, την κρίση, την παρούσα, να την διαχειριστούμε χάρη σε περισσότερη Ευρώπη. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Το συμβόλαιο αυτό, η Σύνοδος Κορυφής θα ασχοληθεί, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, θα πρέπει να ανακτήσουν την δυνατότητα να διαχειριστούν τα, τα κράτη τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν αποφασίζουν πλέον αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το τι συμβαίνει μέσα σε ένα κράτος, αλλά οι 43 μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν μερικές φορές πολύ μεγαλύτερο ΑΕΠ ε, μάλλον ε, κεφάλαιο, η αξία οικονομική, από το ΑΕΠ της Πολωνίας. Άρα είναι ισχυρότεροι οι ε, διοικητές αυτών των ε, επιχειρήσεων, των 43 επιχειρήσεων, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας, Φερρυπίν. Και... Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι μηχανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας προβαίνουν την παραμονή ακόμη ενός Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ σε κρίση και υποβάθμιση κατά μία, δύο, τρεις μονάδες κρατών της ζώνης του ευρώ. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτούς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστονομικής ε, δυνατότητας, ποιοι είναι αυτοί, δεν είναι κάποιοι τυχαίοι, κάποια συμφέροντα εκπρόσωπούν και για κάποιες προτάσεις αξιολόγησης παίρνουν και τη σχετική αμοιβή, το αντίτιμο. Πρέπει λοιπόν να ανακτήσουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το δικαίωμα στη δημοκρατική δράση, στη δημοκρατική διακυβέρνηση. Αυτό μπορούν να το καταφέρουν μόνο αν είναι ενωμένοι. Δεν μπορούν να το καταφέρουν αν ο καθένα κοιτάει σε διαφορετική κατεύθυνση. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει 7,8% του παγκόσμιου πληθυσμού στα 27 κράτη-μέλη της. και έχουμε προβλέψεις δημογραφικές ότι μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια θα έχουμε μόνο 4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δεν θα μπορούμε λοιπόν μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, τις νέες δυνάμεις που αναδύονται, τις ε, νέες οικονομίες που ενισχύονται. Δεν είναι δυνατόν από τη Μεγάλη Γερμανία μέχρι τη πιο μικρή Πάλτα να περιμένουμε, να κατακαιρματιστούμε και να διαλυθούμε. Θα πρέπει μόνο σε μια μεγάλη ένωση και δια, διυπηρωτική αντιπαράθεση να υψώσουμε το ανάστημα, τόσο στο θέμα του περιβάλλοντος όσο και στο θέμα της οικονομίας, της παγκοσμιοποίησης μόνο εάν είμαστε ενωμένοι και αν έχουμε το θάρρος να σταθούμε ως η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου γιατί αυτό είναι η Ευρώπη και μπορεί να στεφθεί με επιτυχία αυτό το μεγάλο εγχείρημα μόνο εάν είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας. γιατί ισχύς εν και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα όχι απλώς φόρος χρηματοπιστωτικό φόρος αλλά φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όταν πουλάω γάλα στο σούπερ μάρκετ πρέπει να πληρώσω φόρο προσθέμενης αξίας. Όταν, Όταν πουλάω χρηματοπιστωτικό προϊόν πρέπει και εκεί πάνω να πληρώνω κάποιο φόρο. Δηλαδή φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Είναι τα δεδομένα όλα επιτάπητος τα βλέπουμε ξεκάθαρα. Και ή θα τα καταφέρουμε με την ενότητα στην Ευρώπη και όχι με το να παίζει παιχνίδια εις βάρος του ενός κράτου το, κράτους στο άλλο και όχι με το να υπάρχουν αντιπαραθέσεις και εντάσεις μεταξύ μας. Μόνο ενωμένοι λοιπόν και για αυτό το λέω διότι η Ευρώπη είναι σε κίνδυνο και πολύ συγκεκριμένο κίνδυνο. Διότι εάν αποτύχει ως υπερεθνικό εγχείρημα η Ευρώπη Εάν καταρρεύσει η Ευρώπη, κυρίε και κύριοι, δεν, δεν καταραίει μόνο μια πολιτική ενότητα. Ξυπνάνε πάλι τα παλαιά δαιμόνια, τα δαιμόνια του 20ου αιώνα, εκείνα που μας έφεραν στο χείλος του γκρεμού. Η διάλυση της Ευρώπης σημαίνει διάλυση και εξαφάνιση μιας πολύ μεγάλης ιδέας.